την ε, κυρία Κάουφμαν πρώτα και το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έναυσμα για αυτή την έκθεση είναι η ανακοίνωση του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα για την αποτελεσματική χρήση ε, τη νομοθετική διαδικασία, το λεγόμενο REFIT. Εν μεταξύ έχει περάσει αρκετό χρόνο χωρί να γίνει τίποτα. Το REFIT υπάρχει το 2012. Είχε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει. Το μεταξύ υπάρχει μια φιλόδοξη ε, διοργανική συμφωνία μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα REFIT ε, έχει κεντρικό ρόλο για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επηρεάσει και τη συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων στην ε, νομοθετική διαδικασία. Ήρθε πλέον η ώρα να συστήσουμε και εμείς και να τοποθετηθεί το σώμα για το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου να εκθέσω κάποιες πτυχές της εκθέσεως ε, που, έχουν, που έχει εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ο Τίμερμανς, ο κύριος Τίμερμανς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλαβε το θέμα αυτό της καλύτερη νομοθέτηση. Ε, και αυτό το κρίνω θετικά γιατί αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε ότι είναι υπερβολική η γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσε σωστά να αλλάξει αυτό. Ιδιαίτερα υπογραμμίζει η έκθεση ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι αν υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη νομοθεσία. Όταν μιλούμε για καλύτερη νομοθεσία πρέπει να μας απασχολεί πάνω απ' όλα η ποιότητα και θα υπενθυμίσω ότι ένας, ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα ε, που αντικαθιστά 28 διαφορετικά νομοθετήματα θα πρέπει να οδηγεί σε λιγότερη γραφειοκρατία και να ενισχύει την ε, κοινή ε, στάση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν έτσι να διασφαλίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά με τρόπο διαφανή και συνεπή προς την νομοθετική διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται στις διαβουλεύσεις να λαμβάνει υπόψη επαρκώς τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα απαιτούνται επίσης όσον αφορά την ενσωμάτωση των διαφόρων στοιχείων και σχολείων που έχει ενσωματώσει στο στην πλατφόρμα Refit ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επευθυνόμενους Πολίτες. Ε, δεν λειτουργεί ακόμη αυτή η πλατφόρμα επαρκώ, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει πω το Κοινοβούλιο θα τη συνοδεύσει ε, και θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αυτή. Επίση, συζητούμε με την έκθεση αυτή ε, να λάβουμε έναν ισχυρότερο και σαφέστερο ρόλο στην ε, νομοθετική διαδικασία. Πώς, από πού ξεκινάει, πώς προκύπτει ένα νομοθέτημα. Αυτά είναι αισθήματα που μας απασχολούν και με την έκθεση καθίσατε σαφές ότι η Επιτροπή για τον κανονιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σε θέση να διατυπώσει δεσμευτική ε, γνωμοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκτελεστικό όργανο, έχει την πολιτική ευθύνη και καλείται να αποφασίσει και αναλόγως να αναλάβει και τις ευθύνες της η αξιολόγηση συνεπειών δεν μπορεί να υποκαταστήσει καμία πολιτική απόφαση. Όσον αφορά την εμπλοκή και των κοινωνικών εταίρων, Βεβαίω πρέπει να ισχύει η αρχή τη, αυτονομίας τους, η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων δηλαδή. Οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει θα υποφεληθούν ιδιαίτερω από την επίσταση τη γραφειοκρατίας, αποτελούν, όπω ξέρουμε, την αρχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Ταυτόχρονα όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επιχείρηση. Η καλύτερη νομοθεσία δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο με όρους ε, επιχειρηματικούς, δηλαδή κόστους και ωφέλους, με οικονομικούς όρους. Δεν πρέπει ε, στη διαδικασία αυτή να αμφισβητούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων, επί παραδείγματι, ή η εσωτερική αγορά σε κατακαιρματισμό με διαφορετικές ρυθμίσεις αναλόγως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ρίφιτ για να ολοκληρώνω Πρόεδρε, θα συνεχίσει να μας απασχολεί, θα το παρακολουθούμε με ιδιαίτερη έμφαση. Θέλω να ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο Επιτροπής και βεβαίως ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ με το σύστημα αυτών των σύντομων παρουσιάσεων ε, περνούμε κατευθείαν στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΕΡ και τη συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Κυρία Νίβλερ πρώτα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή εισηγήτρια. Θέλω πολύ στήμα να πω ότι το ΡΕΦΙΤ είναι ένα καλό πρόγραμμα, είναι ευπρόσδεκτο το να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποσύρει συγκεκριμένε προτάσει. Είναι κάτι το οποίο έχει προεξαγγείλει και η Επιτροπή Γιουνκέρ, ε, ε, το θεωρούμε ευπρόσδεκτο λοιπόν. Θέλω απλώ να αναφερθώ στο θέμα των συνεπειών τη νομοθετική διαδικασία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλέ φορέ επιμένουμε και εδώ και χρόνια ζητούμε όταν γίνονται προτάσει για τροποποίηση που έρχονται στο Κοινοβούλιο για να γίνουν ε, νομοθέτημα να υπάρχει μια πλήρη αξιολόγηση των συνεπειών τη αγωγή αυτή τη νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στην υπόθεση αυτή. Υπάρχει μια επιτροπή ή υποεπιτροπή κανονιστικού ελέγχου εμείς ζητούμε να ε, συσταθεί ένα ανεξάρτητο Συμβουλίο Αξιολόγησης Κανονιστικών Συνοπιών. Αντίστοιχα υπάρχουν τέτοια όργανα και στη Γερμανία, τι κατοχώρες, στη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με, αυτό το, με αυτή την επιτροπή, υποεπιτροπή κανονιστικού ελέγχου κάνει ένα βήμα προς τα πίσω και θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση ανεξάρτητου οργάνου. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Νεγκρέσκου, ένα λεπτό. ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το έγγραφο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο με στα πλαίσια του REFIT. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο με βάση αρμοδιότητες της πρώτης αντιπροέδρου της Επιτροπής. Θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη με τον πολίτη. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Επίσης, θα πρέπει να μιλάμε για 12 εβδομάδες διαβούλευσης με τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την νομοθεσία αλλά και οι πολίτες να πληροφορούνται όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νεγρέσκου και τώρα ο κύριος Μαριάς κύριε πρόεδρε σαν καθηγητή θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πανεπιστήμιο τη Κρήτη, έδινα πάντα και συνεχίζω να δίνω μεγάλη σημασία στο ρόλο τη επιτροπής διότι η επιτροπή είναι ο θεματοφύλακα τη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. η επιτροπή διαθέτει τα εργαλεία εκείνα που τη επιτρέπουν να κρίνει την αποδοτικότητα και καταλληλότητα του νομοθετικού έργου που παράγουν οι θεσμοί. τα εργαλεία αυτά πρέπει βεβαίω να βελτιωθούν. Όμω η επιτροπή δεν πράττει το ίδιο κυρία γιουρόβα ω μέλο τη τρόικα στην ελλάδα διότι εκεί αναδεικνύεται η σύγκρουση συμφερόντων. εκεί η επιτροπή ενεργεί καθαρά ως εκπρόσωπος των δανειστών. και θα σας φέρω ένα παράδειγμα αυτό το διάστημα πιέζει η τρόικα στην ελλάδα να ληφθούν μέτρα για το συνταξιοδοτικό για το ύψος των συντάξεων για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και εγώ ρωτώ με ποια αρμοδιότητα παρεμβαίνει η επιτροπή. τα θέματα των συντάξεων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών το ίδιο κάνετε και με τη φορομπηχτική πολιτική που επιβάλλεται στην ελλάδα. επομένως εκεί ως μέλος της τρόικας εκφεύγετε των αρμοδιοτήτων σας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική. Ο κύριος Τίμερμανς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αναφέρθηκε πάνω από μια φορά σε αυτό το ζήτημα. Όμως τι κάνουμε πραγματικά για να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και για να κάνουμε τα πράγματα πιο σαφή ως προς την νομοθεσία. Να γίνεται δηλαδή και η νομοθεσία πιο σαφής και κατανοητή και από τους ε, πολίτες ιδίως όσους που είναι κατά κάποιον τρόπο πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αναφέρομαι στις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και τι συμβαίνει με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χιλιάδες διαφορετικούς κανόνες, ε, διατάξεις μπορεί να είναι απαραίτητε, αλλά δεν είναι σαφεί. Δεν τι κατανοεί ο κόσμο που πρέπει να τι χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να απλουστευτούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νόβα Κοφένα λεπτό. <clears throat> Ευχαριστώ. Το Refit είχε σχεδιαστεί ω ε, ένα τείχο προστασία το 2012. Το πρόγραμμα έχει ε, πολύ μεγάλη επιτυχία με πάνω από 200 δράσει και το καθεξής. Όμω δεν καλύπτει τα πάντα. Θέλουμε να προσθέσουμε τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Όμω, το βασικό έγγραφο δεν είναι και τόσο απλό και φιλικό προ το χρήστη όσο θα θέλαμε. Το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 έχει 40 ενέργειε και πρωτοβουλίε REFIT, αλλά καμία δεν προβλέπει ε, περιορισμό του διοικητικού ε, δικαίου και αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα Έχουμε πάνω από 250 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για επιμέρους ε, πρωτοβουλίες που ουσιαστικά θα χαθούν μέσα στις γραφειοκρατικές ε, διόδους. Το 95% των ευρωβουλευτών υπερψηφίζουν διατάξει για τον περιορισμό ε, τη γραφειοκρατίας. Όμω όλα αυτά δεν υπάρχουν μέσα στο ψήφισμα. Στηρίζω την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Αυτό είναι το θέμα. Äh, äh, Ευχαριστώ η Επιτροπή. Η Επιτροπή Γιώργο έχει το λόγο. Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάουφμαν για την έκθεση για το ReFit. Τα αποτελέσματα αποτελούν μία ενθάρρυνση στην εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό για μένα προσωπικά ο ε, ευρωπαϊκός νόμος θα είναι, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός, να μην είναι τόσο δαπανηρός και να μπορεί να εφαρμοστεί στα, σωστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλα τα θεσμικά όργανα. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ε, νέων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κόπωσης που μας απασχολεί πολύ συχνά. Υπάρχει μια διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση που εγκρίνεται το Μάρτιο. Η έκθεση όμως αυτή είναι προγενέστερη της συμφωνίας. Γι' αυτό πολλά από τα θέματα που φύγει έχουν επιληθεί. Στο μεταξύ η Επιτροπή ε, έγκρινε στις 19 Μαΐου 2015 το πακέτο για, την ε, καλύτερη, για το καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ και άλλους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Υπήρχαν πολλά μέτρα, δηλαδή ένα νέο συμβούλιο ε, ελέγχου το οποίο έχει συσταθεί και αποτελείται από ε, εμπειρογνώμονες εκτός κομισιών και γίνεται και μία εκ των υστέρων αξιολόγηση. Επίσης υπάρχουν τα μέσα για να μπορούμε να εφαρμόσουμε την ε, καλύτερη ε, ρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή τον έλεγχο της αξιολογήσης και το νομοθετικό έργο και τσεπτό στο περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά που έχει εγκριθεί ένα τέτοιο έγγραφο στην Επιτροπή. Έχουμε μια τέτοια νέα πλατφόρμα του ReFit. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα τον Ιανουάριο και ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Η νέα Διαθεσμική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθέτηση ε, αφορά και εμπεριέχει πολλά επιτεύγματα για κατεξιοδότηση πράξης και εκτελεστικές πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε αυτή τη συζήτηση μεταξύ των από κοινού νομοθετών. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο των κατεξιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων πριν εκδοθούν. Επίσης χρειάζεται ε, ένα διαχρονικό πρόγραμμα όπου προβλέπεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων μέσα στα πλαίσια των ε, πολιετών προγραμμάτων και η προετοιμασία των ε, χαρτοφυλακίων ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο του REFIT θα δούμε πώς θα αποτιμάται το περιεχόμενο στο μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την εφαρμογή του. Το ε, πρόγραμμα ε, καταλληλότητας του REFIT θα λάβει υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία και θα μειώσει τον ε, ρυθμιστικό φόρτο χωρίς να αποδυναμώσει περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους ως προς την διαφάνεια. Θα πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού για κοινέ πλατφόρμες, για τις κατεξιοδότηση πράξης και τη δυνατότητα συνομοθέτησης έτσι ώστε και το κοινό να μπορεί να ελέγχει τις νομοθετικές πράξεις. Μετά την επίσημη έγκριση, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να γίνει έγκαιρη εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη νομοθέτηση για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό τη διάταξη. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό θέλετε. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα διάκρισης. Δύο φορές ε, θέλαμε να προσελκύσουμε την προσοχή σας στο Catch the Eye, αλλά δεν μας λάβετε ε, υπόψη και στις δύο συζητήσεις. Ε, Όταν έχουμε 9, 10, μερικέ φορέ και 18, 19 ε, αιτήματα για catch the eye, δεν μπορούν να λάβουν όλες οι ομάδες ε, το λόγο. Οι μεγαλύτεροι ίσως να πάρουν μια-δυο φορές το λόγο και οι μικρότερες μόνο μία, αλλά δεν πρόκειται για διάκριση, πρόκειται προς η κατανομή του χρόνου. Και περνώ στο θέμα